So, uh, Αγαπητοί συναδελφοί, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στην απογευματινή συνεδρίαση. Θα πραγματοποιήσουμε κοινή συζήτηση ε, με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σχέση με τις χώρες Μαγκρέμπ. Ιδιαίτερα χαίρομαι για αυτή την ευκαιρία. Και βέβαια για το γεγονό ότι συμπροεδρεύω με την πρόεδρο τη αντιπροσωπεία για το Μαγκρέπ, την κυρία Γιάλα Σάντερ. Βέβαια η έκτο έχει πολύ μεγάλη σημασία και μα ενδιαφέρει πάρα πολύ, όπω και η Λιβύη, για την οποία έχουμε ετοιμάσει μία ε, επίσκεψη στο βαθμό που δεν έχουμε προσωπικές ε, ε, πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνούμε με τους εκπροσώπους που επισκέπτονται τη χώρα και έτσι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή, το τι γίνεται αυτή η κοινή συνεδρίωση. Και βέβαια η ενημέρωση για το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της 27 Ιανουαρίου που αφορά συγκεκριμένα την ε, Λιβύη θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Καλώς ήρθατε, φτάσατε ίσα ίσα στην ώρα σας και σας καλωσορίζω κύριε Βίνσεντ Πικί και κύριε Αμρόζη. Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης έχουμε προσκαλέσει και την Υπατή που δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει, θα μας ε, ε, έχει αποστείλει όμως και θα το βρείτε στα έγγραφα της συνεδρίασης, στα ενημερωτικά της Δελτία. Δίνω το λόγο στην κυρία Γιάλα Σέντερ για να μας κάνει την παρουσίαση. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις, ε, τα βαθές συλληπιτήρια για τις οικογένειες ε, των θυμάτων στη Λιβύη. θυμάτων των τρομοκρατικής επίθεσης και βέβαια όλων των εργαζομένων στον χώρο της υγείας και της περίθαλψης. Ε, ασφαλώς και όλες οι ευχές μας και προσευχές μας ε, πάνε σε αυτό, στην ειρήνη και στην ασφάλεια στη Λιβύη, ώστε να μπορούν να ζουν ε, με ασφάλεια οι πολίτες. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, το ξέρουμε, αλλά αυτές είναι οι προσπάθειές μας και θέλουμε ως Ένωση να εκδηλώσουμε την αλληλεγγύη μας με τα συλληπιτήριά μας προς τα θύματα και τους οικείους τους εκ μέρους της Μαγκρέμπ Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως την Επιτροπή σας για αυτή την κοινή συνεδρίαση. Για, τις, ε, για την ευκαιρία αυτή και βέβαια και τους εκπροσώπους, ε, τον κύριο Πικέ που είναι εδώ κοντά μας, για να μας ενημερώσει για την εξέλιξη των συνομιλιών και τα κύρια προβλήματα όπως τα διαβάζει. Η αρχή που εκπροσωπεί και τον κύριο βέβαια Αμπρόζη. Στις 22 λοιπόν Ιανουαρίου το Συμβούλιο πραγματοποίησε συζήτηση για τη Λιβύη για να εξετάσει την κατάσταση στη χώρα και ο εκπρόσωπος των Αθηνών μου Σαλαμέ έκανε μια σύνοψη της κατάστασης, πολιτικές προόδους και δυνατότητες για εξασφάλιση ενός νέου συντάγματος με τις, προσ... με τις προσεχείς εκλογές. Φυσικά, του δόθηκε αμέριστη υποστήριξη από τους Υπουργούς Εξωτερικών στις προσπάθειες του αυτές, που όπως είπα στόχο έχουν την επανασυμφιλίωση και ειρήνευση στη χώρα. Επίσης συζήτησαν τη σημασία της ε, παρουσίας και δέσμευσης της ε, στράτευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη, οι Υπουργοί. με στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών της, ε, του Οργανισμού Εθνών και συγκεκριμένα των διάφορων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ε, μετανάστευσης, της διαχείρισης μεταναστευτικών ροών κτλ. Οι Υπουργοί των Εξωτερικών υπογράμμισαν επίσης ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τις χώρες προελεύσεως των μεταναστευτικών ροών, ιδιαίτερως εκείνων ε, της ε, ζώνης του Σαχέλ και καθώς η συνεδρίαση που διεξέχουμε τώρα είναι κοινή με τη ΛΥΜΠΕ περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τους προσκεκλημένους μας που θα μας δώσουν τις πιο πρόσφατες ε, πληροφορίες σε σχέση με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην συνεργασία με τον ΟΗΕ και μια και είμαστε και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, πληροφορίες και για την κατάσταση των μεταναστών που βρίσκονται στη Λιβύη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριες ε, Πρόεδροι που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την προσέγγισή μας όσον αφορά τη Λιβύη. Έχω ένα κείμενο το οποίο θα χρησιμοποιήσω. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη των περασμένων δύο ημερών δείχνουν πόσο άχρηστα είναι τα έτοιμα κείμενα. Πριν από δέκα μέρες, Είχαμε τι συγκρούσει στο μόνο λειτουργικό Διεθνέ αεροδρόμιο της Τρίπολη. Πολλοί κόσμος έχασαν τη ζωή του και άμαχοι. Διεκόπη η ενέργεια κυκλοφορία για σχεδόν μια εβδομάδα. Παρεμποδίστηκε και μια ευρωπαϊκή ε, κοινή δράση με το Ηνωμένα Έθνη ε, και την Αφρικανική Ένωση που μετέβαινε εκεί πριν από δύο μέρες στη Βενγάζη Είχαμε μια ε, φρικτή ε, διπλή ε, τρομοκρατική επίθεση με βόμβα, βομβιστική επίθεση με αυτοκίνητα. Πολλοί κόσμος έχασε τη ζωή του, πολλοί τραυματίστηκαν, επηρεάστηκε πολύ σημαντικά η σταθερότητα και το περιβάλλον ασφάλειας στη χώρα. Χθες λάβαμε αποτρόπες εκθέσεις για έξω δικαστικές ε, δολοφονίες 10 ατόμων. Κανείς δεν γνωρίζει ποιοι ακριβώς σκοτώθηκαν. Με συνοπτικές διαδικασίες ε, έγιναν ε, οι εκτελέσεις από έναν από τους διοικητές του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, τον διοικητή Χάφτερ, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα πολέμου ε, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας. Όλα φυσικά αυτά παρεμποδίζουν ε, ε, και διάφορες δράσεις άλλες δείχνει πόσο δύσκολο είναι το κλίμα στη Λιβύη σε τι κίνδυνο βρίσκονται οι δυνάμεις ασφαλείας ε, και πόσο υπονομεύεται το περιβάλλον ασφαλείας και δείχνει επίση σε ποιο βαθμό η Λιβύη και ο κόσμος ολόκληρος ε, χρειάζονται μια πολιτική λύση για αυτή την πολιτική κρίση. Ω εισαγωγή στη σύντομη μου παρουσίαση ε, των όσων ε, έλαβαν χώρα τη Δευτέρα στην ε, συνάντηση εξωτερικών υποθέσεων με τη συμμετοχή του ε, είπα το εκπροσώπου Χασάν Σαλαμέη από τα Ηνωμένα Έθνη με μια πλήρη ενημέρωση εκ μέρους τους στους Υπουργούς Εξωτερικών και που ακολουθήθηκε από μια πολύ καλή συζήτηση. Το επίκεντρο της συζήτησης ήταν φυσικά μία από τις δύο βασικές ε, οδούς ε, όπου εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λιβύη, ε, η πολιτική οδός. που υποστηρίζει το σχέδιο δράση των ΗΕ, το οποίο παρουσίασε ο κ. Σαλαμάη πέρυσι, το Σεπτέμβριο λίγο μετά από τον ε, διορισμό του. Ε, κάποια χαρακτηριστικά του σχεδίου αυτού, από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η πρόθεση διεξαγωγής εκλογών στη Λιβύη, προεδρικών εκλογών, καθώς και κοινοβουλευτικών, εξαιρετικά δύσκολο έργο στο περιβάλλον της Λιβύης, ειδικότερα επειδή αυτή τη στιγμή η εκλογική βάση ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει σύνταγμα που να διέπει το ρόλο ενός Προέδρου, που να θεσπίσει το ρόλο Προέδρου και δεν υπάρχουν και νομικές διευθετήσεις ε, για το πώς ε, ε, ένας Πρόεδρος θα ε, λειτουργούσε μαζί με μια κυβέρνηση και ένα κοινοβούλιο. Για να πραγματοποιηθούν λοιπόν τέτοιε εκλογέ πρέπει να γίνουν γίνει πολλέ προπαρασκευαστικέ ε, ε, νομικέ εργασίε. Το καλό είναι ότι έχει ξεκινήσει η εγγραφή των ψηφοφόρων και ο, ο εκπρόσωπος των ΗΕ έδειξε αισιοδοξία ότι όλα αυτά θα γίνουν σε εύλογο χρόνο πριν από την ε, προθεσμία. Κάτι άλλο σημαντικό για τη διεξαγωγή εκλογών και για τη θέσπιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου είναι η οργάνωση μιας ε, εθνικής διάσκεψης για την οποία ο κ. θέλει να υπάρχει συμμετοχή πολλών διαφορετικών ενδιαφερομένων από όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και φιλετικής ζωής της Λιβύης. Κύριος σκοπός αυτής της διάσκεψης θα είναι η ε, δημιουργία μιας ευρείας πολιτικής συνένεσης η οποία θα διασφαλίζει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα γίνει δεκτό από την πολιτική τάξη. Η οργάνωση αυτής της εθνικής διάσκεψης φυσικά δεν είναι κάτι απλό. Γι' αυτό το λόγο, κύριο Σαλαμέ, θα ακολουθήσει μια βηματική προσέγγιση, ξεκινώντας από διάφορες ε, μικρές ε, διασκέψεις για την προετοιμασία της η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εκπρόσωπος, είπατε εκπρόσωπος έχουν αναφέρει ότι θέλουν να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία διότι μόνο με εκλογές στη χώρα αυτή βάσει ενός συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου και ιδανικά με την υθέτηση ενός συντάγματος ε, ε, θα υπάρχει μια αποδεκτή νομική βάση. Ε, εφόσον υπάρχει μια αποδεκτή νομική βάση για τις εκλογές μόνο έτσι μπορεί να καθιερωθεί μια βιώσιμη πολιτική λύση στη, για τη σημερινή πολιτική κρίση. Αυτή είναι μια σημαντική οδός. Η δεύτερη σημαντική οδός ε, που συζητήσαμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δευτέρα αφορούσε την οικονομική πλευρά των πραγμάτων όπου η εικόνα είναι λίγο σύνθετη. Από τη μία πλευρά, σε μακροοικονομικό επίπεδο, τα αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, οπότε και τα σχετικά εισοδήματα. Η παραγωγή της Λιβύης ε, υπήρξε σταθερή πάνω από ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, οπότε τα ταμεία της Κεντρικής Τράπεζας γεμίζουν ε, σταδιακά και υπάρχει χρήμα για διάφορες δαπάνες. Ωστόσο δεν δαπανάται χρήμα επαρκώς, ούτε σωστά. Πολλά από αυτά φεύγουν σε μισθούς, σε κρατικό προσωπικό, προσωπικό ασφαλείας, ε, ορισμένοι από τους οποίους ε, λειτουργούν και κάπως άτυπα και ελάχιστα ουσιαστικά χρήματα πηγαίνουν στα Υπουργεία, στις δημόσιες που απαιτούν χρηματοδότηση για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Παρά λοιπόν την καλή μακροοικονομική κατάσταση ε, και, και τη σταθερότητα στις συνταγματικές ισοτιμίες ε, υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος. Τα καλά νέα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα συμμετέχει στον επωνομαζόμενο οικονομικό διάλογο που διεξάγεται εδώ και κάποιο καιρό στην ε, Λιβύη, χωρίς την Ευρώπη, αλλά από την περασμένη εβδομάδα συμμετέχουμε και εμείς και με μεγάλη μας χαρά θα δώσουμε και εμείς ε, τη δική μας συμβολή στον πολιτικό αυτό προβληματισμό, του οποίου φυσικά έχουν οι ίδιοι Λιβύοι. Αυτά ε, στην πολιτική και την οικονομική οδό. Τελευταίο θέμα η μετανάστευση που φυσικά συνεχίζει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, πρώτη προτεραιότητα ε, όχι μόνο για το UNHCR αλλά και για τον πρόσωπο Ουσιαστικά το 2017, και θα το συζητήσουμε πιο λεπτομερώς, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, λιγότερες αφήξεις στις ευρωπαϊκές ακτές, ε, άτυπων μεταναστών, ε, λιγότερη θάνατη στη θάλασσα, γεγονός φυσικά που αποτελεί μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα, ε, περισσότεροι διασωθέντες, από τη θάλασσα και περισσότερος κόσμος έχει ε, επιστραφεί από τη Λιβύα στις χώρες καταγωγής τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος ε, στο οποίο συνεργαζόμαστε και εμείς με τον ε, Διεθνή Οργανισμό Μεταναστευση και την UNHCR για τις εθελοντικές επιστροφές. Έχουν επιληθεί όλα, όχι φυσικά, αλλά το γεγονός είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός άτυπων μεταναστών εντός της Λιβύης, 600.000 περίπου. και ενδεχόμενη ε, δημιουργία προβλημάτων λόγω αυτών. Εξακολουθούν να υπάρχουν και πολλοί άτυποι μετανάστες οι οποίοι κρατούνται σε κέντρα κράτησης που λειτουργούν ε, υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Ορισμένα κέντρα κράτηση ε, ε, τα διαχειρίζονται άτυπες ομάδες που δεν ελέγχει κανένας ουσιαστικά, αυτό ελέγχονται με τη συνέπεια σημαντικά ανθρωπιστικά ζητήματα, ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και γι' αυτό το λόγο είπατε εκπρόσωπος αποφάσισε να συζητήσει ε, μαζί με το Ηνωμένα Έθνη και την Αφρικανική Ένωση ώστε να, ενταθούν να ενταθεί η βοήθεια για τις εθελοντικές επιστροφές όσον αφορά τους κρατουμένους στα κέντρα αυτά με στόχο να πείσουμε τη λιβική πλευρά να διακόψει αυτή την πρακτική της εγκληματικής κράτησης των άτυπων μεταναστών. Αυτός είναι ο στόχος. Ταυτόχρονα φυσικά θα αρκεστούμε σε μια ενδιάμεση λύση. δημιουργίας ε, κέντρων κράτησης που να τηρούν τις ανθρωπιστικές συνθήκες. Κάτι άλλο νέο ήταν η δημιουργία της Task Force μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης 29 Νοεμβρίου στο Αμπιτζάν. Έγινε μια συνάντηση στις Βρυξέλλες στις 14 Δεκεμβρίου ε, για τον προγραμματισμό των εργασιών. Με βασικό στοιχείο το πρόγραμμα ε, υποβοήθησης, ε, βοήθηση, αρρωγής προς την εθελοντική επιστροφή ε, ένα πρόγραμμα στο οποίο θέλουμε και τη συμμετοχή των λιβικών αρχών, ε, κάτι φυσικά που ισχύει διαρκώς, αλλά είχαμε ελπίσει να γίνει όλο αυτό στο πλαίσιο μιας κοινή αποστολής με τα Ηνωμένα Έθνη και με τους συναδέλφους από την Αφρικανική Ένωση. Αυτή την εβδομάδα, 22 του μήνα, την περασμένη Δευτέρα ουσιαστικά, διακόπη αποστολή ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων στο αεροδρόμιο. Αναβλήθηκε δηλαδή η αποστολή για το μέλλον με στόχο τώρα να κινητοποιηθεί κάπου στις 20 ε, Φεβρουαρίου. Αυτά, έτσι έχει η σημερινή κατάσταση. Η ουσία είναι ότι σε όλους τους τομείς ε, χρειάζεται συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, πλήρης υποστήριξη για την πολιτική διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών και πολύ στενή ε, συνεργασία με τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε ε, κύριε Βικέ ε, για όλες αυτές τις ε, λεπτομερείς πληροφορίες. Ο κύριος Αμπρός έχει τώρα το λόγο. Thank uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και καλησπέρα σε όλους. Πολύ σύντομα. Να σας ενημερώσω ως προς τη δική μας οπτική γωνία σε σχέση με το τι συμβαίνει στη Λιβύη και το τι προσπαθούμε εμείς να κάνουμε Αποκινούμε τους εταίρους μας ειδικότερα βέβαια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια κράτη-μέλη στιγμά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά βέβαια έχοντας ε, κατά νου την γενικότερη ε, κατάσταση την πολιτική ασφαλείας η οποία βέβαια ουσιαστικά αποτελεί και το γενικό υπόβαθρο και έχει και το μέγιστο αντίκτυπο στα όσα προσπαθούν να κάνουν όλοι οι εταιρείε εκεί και οι υπηρεσίε των Ηνωμένων ε, επί τόπου στο πλαίσιο δηλαδή της ε, ανταπόκρισης στις αρμοδιότητες του στην εντολή τους. Ουσιαστικά τρεις κατηγορίες ανθρώπων εμείς ε, έχουμε ως ομάδες στόχους των εργασιών μας. Τρεις κατηγορίες οι οποίες σχετίζονται βέβαια στενά μεταξύ τους. Καταρχήν οι εσωτερικά ιδιωγμένοι ε, πολίτες της ε, Λιβύας, ε, γύρω στους 80.000 σε αυτή τη φάση έχουμε εσωτερικά, εσωτερικά εκδιωγμένους. Ένας αριθμός όμως ο οποίος ευτυχώς μειώνεται. Όχι βέβαια με πολύ μεγάλους αριθμούς αλλά στάθερα κάτω στους τελευταίους Λιβύοι πολίτες δηλαδή της Λιβύης αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους έτσι ώστε να βοηθήσουν στην ανοικοδόμησή τους. Ανοικοδόμησή της και προφανώς αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία ατόμων τα οποία προσπαθούμε να υποστηρίξουμε, δηλαδή την επιστροφή τους στην πατρίδα τους και την ε, διασφάλιση της δυνατότητας να παραμείνουν εκεί και να ξεκινήσουν μία ε, σε κάποιο βαθμό αξιοπρεπή ε, διαβίωση εκεί, υποστηρίζοντας τη σταθεροποίηση της χώρας και την πολιτική διαδικασία που μόλις τώρα περιγράφηκε. Η τρίτη κατηγορία ατόμων είναι φυσικά οι μετανάστες. έχουμε καταχωρήσει γύρω στους 620.000 ε, μετανάστες επισήμως, αλλά βέβαια η κατάσταση στη χώρα είναι τέτοια που να μην μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις περιοχές της χώρας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι πράγματι 620.000 άτομα είναι ο συνολικός αριθμός. Ε, οι εκτιμήσεις μας ε, ανέρχονται σε 800.000, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Εκεί περίπου λοιπόν κυμαίνονται οι αριθμοί των εκτιμήσεών μας σε ό,τι αφορά τους μετανάστες στη Λιβύη, οι οποίοι είναι διασπαρμένοι σε ολόκληρη τη χώρα και ένα μεγάλο τμήμα τους, ε, γύρω στο 50% με βάση τις ε, πληροφορίες που έχουμε και τις συνεντεύξεις που έχουμε λάβει, είχαν ως κύρια πρόθεσή τους όταν εγκατέλειψαν τη χώρα τους ε, τη Λιβύη για να εργαστούν. Γιατί παραδοσιακά αποτελεί ακριβώ χώρα προορισμού τη μετανάστευση για λόγου τη εργασία ε, και ε, σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζεται και οικονομικά από τέτοιου ε, μετανάστε εργαζόμενου. Άρα λοιπόν, όσο και να ακούγεται ενδεχομένω απίστευτο, πράγματι αυτό είναι ο στόχο πολλών μεταναστών που βρίσκονται στη Λιβύη, δηλαδή να εργαστούν εκεί. Η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών που βρίσκονται στη Λιβύη δεν έχουν ε, αρχικά το στόχο λοιπόν να μεταβούν στην Ευρώπη. Αυτός ε, καθίσταται ένας δευτερεύον, αν θέλετε, ένας δεύτερος στόχος όταν τελικά δεν καταφέρνουν να βρουν την εργασία ή να κάνουν αυτό που ήθελαν στη Λιβύη. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντικό σε πολιτικό επίπεδο να διασφαλίσουμε την ε, σταθεροποίηση σε διάφορες κοινότητες της Λιβύης γιατί με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα μειώσουμε ε, τον αριθμό αυτών των μεταναστών οι οποίοι ως δεύτερη επιλογή αν θέλετε επιλέγουν να προσπαθήσουν να μεταβούν στην Ευρώπη. Από εκεί και μετά υπάρχουν και κάποιες καλές ειδήσει. Ε, ήδη την ανέφερα. Είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των εσωτερικά εκδιωγμένων στη Λιβύη, ο οποίος τελικά μεταβαίνει στην πατρίδα του και παραμένει εκεί, ε, μειώνεται. Με σταθερούς ρυθμούς που αυτό σημαίνει βέβαια ότι η χώρα καθίσταται σταδιακά αρκούντο σταθερή έτσι ώστε οι εσωτερικά ιδιωμένοι να επιστρέψουν ε, στην, ε, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και πρόκειται για μια διαδικασία βέβαια η οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί. Η δεύτερη θετική είδηση είναι αυτό που ήδη ακούσαμε ότι ο αριθμός των ατόμων που διασύρουν τη Μεσόγειο από τη Λιβύη με προορισμό την Ευρώπη επίσης μειώνεται στους τελευταίους ε, μήνες. Αλλά βέβαια αυτό περιλαμβάνει και μια προβληματική διάσταση γιατί ο πλήρης σεβασμός των ε, τεμελιωδών δικαιωμάτων αυτών των μεταναστών στη Λιβύη δεν είναι πλήρως εγγυημένος. Οπότε δηλαδή έχουμε μια θετική πτυχή που είναι ο μειωμένος αριθμός των αφήξεων και κατά συνέπεια και των θανάτων στη Μεσόγειο, δηλαδή σώνουμε περισσότερες ε, ζωές αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε την αρνητική διάσταση, το γεγονός δηλαδή ότι οι συνθήκες ε, διαβίωσης ε, δεν είναι κατάλληλε στη Λιβύη και δεν υπάρχει και ο υπαρκή σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτιώσεων και ακριβώ σε αυτό το τομέα θα πρέπει να εργαστούμε παραπάνω και να συνεργαστούμε με τι αρμόδιε αρχέ έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συμμόρφωσή τους με τι θεμελιώδει αρχέ ε, και μεταχείριση των μεταναστών, αλλά γενικότερα όλων των πολιτών. Και εδώ περνάω στο ζήτημα των α, κέντρων κράτησης, ε, που αποτέλεσαν βέβαια το αντικείμενο α, ε, ε, της συμφωνίας που συνήθισε το Αμπιτζάν με την Αφρικανική Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Αποφασίστηκε λοιπόν να αυξηθεί ο αριθμός των πλούσιων επιστροφών από τα κέντρα κράτησης έτσι ώστε να μειωθεί και ο γενικός πληθυσμός σε αυτά τα κέντρα κράτησης με αποτέλεσμα να βελτιωθούν έστω και εν μέρη οι συνθήκες διαβίωσης σε αυτά τα κέντρα κράτησης. Νομίζω πως όλοι είδαμε σε δελτία ειδήσεων, σε βίντεο του CNN και αλλού με πολύ γραφειρό τρόπο να το, το ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν ε, στα κέντρα κράτησης ε, και εγώ ε, έχω, εργάζομαι σε αυτό το τομέα εδώ και 30 χρόνια έχω επισκεφτεί κάθε είδου καταβλισμού προσφύγων, κέντρα κράτηση, εσωτερικά εκδιωγμένων και ούτω καθεξής, αλλά πραγματικά σπανιότατα έχω δει μια τόσο άσχημη κατάσταση. Δεν μπορείτε δηλαδή να φανταστείτε τι συμβαίνει. Δηλαδή φανταστείτε ένα κέντρο κράτησης ε, που προορίζεται για 400 άτομα αλλά μέσα διαβιούν 1000-1200 άτομα και υπάρχουν μόνο τέσσερις τουαλέτες για όλα αυτά τα άτομα. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν τι συμβαίνει. Ο στόχος λοιπόν της συμφωνίας είναι να μειωθεί λίγο ο αριθμός των όσων διαβιούν στα κέντρα κράτησης αλλά φυσικά αυτό προϋπέθεται μία απόφαση ε, από την πλευρά της κυβέρνησης της Λιβύης να σταματήσουν να οργανώνουν με αυτόν τον τρόπο ε, τα κέντρα κράτηση, δηλαδή το πώ καταλήγει κανεί στα κέντρα κράτηση. Αλλά δυστυχώ δεν συμφώνησε να υπογράψει με τέτοια συμφωνία ε, ω προ την αλλαγή του συστήματο η Λιβύη. Άρα λοιπόν παρότι μειώνεται ο αριθμό λόγω ακριβώ τη αύξηση των επιστροφών, υπάρχει ο κίνδυνο να αυξηθεί εκ νέου ο αριθμό στα κέντρα κράτηση λόγω ε, του ίδιου συστήματο που οδηγεί εκεί τα άτομα ε, όταν είχε συνηθίσει σχετική συμφωνία, λόγω των, ε, των μαχών και στην Σαββάτα είχε αυξηθεί ο αριθμός ε, των παραμένοντων σε αυτά τα κέντρα κράτησης στου 20.000, ενώ ότι σήμερα ο αριθμός των κρατούμενων σε αυτά τα κέντρα κράτησης είναι γύρω στους 8.000. Αυτό αποτελεί μία ένδειξη στα κέντρα κράτηση σε κάποιο βαθμό και εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για, τον, για την επιστροφή των διαμένοντων στα κέντρα κράτησης το ταχύτερο δυνατό. Ε, βέβαια, η εταιρική σχέση σε ό,τι αφορά αυτές τις επιστροφές από τη Λιβύη ε, δεν αφορά μόνο τη σύφτη της διαδικασίας αλλά και ένα ιδιαίτερα δύσκολο τμήμα. Γιατί η επανένταξη ατόμων ούτως ή άλλως ως ε, εγχείρημα είναι κάτι το δύσκολο, αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε και με πολύ υψηλότερους αριθμούς από αυτούς που αναμέναμε στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Ε, δηλαδή, για 6.000 ε, και τώρα έχουμε φτάσει σε επιστροφές πάνω από 19.000 ατόμων, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η αύξηση των επιστροφών. Αλλά βέβαια είναι θετικό το αποτέλεσμα, ότι δηλαδή πράγματι μειώνεται η δυστυχία όλων αυτών των ανθρώπων, επιστρέφουν, επανεντάσσονται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολη αυτή η συνεργασία. Και χρειάζεται να βελτιωθεί περαιτέρω. Και... Κάτι τελευταίο. Και από εκεί και μετά βέβαια είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ε, ένας ακόμα σημαντικός τομέας των εργασιών μας είναι της Λιβύης ιστορικά και παραδοσιακά αποτέλεσε ένα από τους κύριους τομείς της Λιβύης που επηρεάζει την σταθερότητα ή την αστάθεια που επικρατεί στη χώρα. Άρα λοιπόν ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να επιτύχουμε περισσότερη κοινωνική συνοχή και σταθεροποίηση και συνεργασία μεταξύ των ε, κατατόπους ηγέτες Λιβύης. Ε, ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα ε, που καθιστά δηλαδή αυτή την περιοχή τόσο σημαντική είναι το γεγονό ότι πολλοί εσωτερικά εκδιωγμένοι επιστρέφουν ακριβώ εκεί, στην Νότια Λιβύη. Άρα λοιπόν με την βελτίωση της σταθερότητας σε αυτή την περιοχή, διασφαλίζουμε το να παραμείνουν εκεί όσοι επιστρέφουν και κινούνται ε, προς βορρά. Άρα λοιπόν, όσο περισσότερη σταθερότητα έχουμε σε αυτή την περιοχή, τόσο λιγότερες οι πιθανότητες εν λόγω μετανάστες να συνεχίσουν αυτό το ταξίδι τους ε, προς βορρά, φτάνοντας σε κάποια φάση ενδεχομένως ε, στα δίκτυα των το προσωπικό μας ε, το οποίο δρεύει στην Σάβα, σε μία από τις πόλεις ε, ε, της ενότιας Λιβύης είχε ένα μέρος του το οποίο το τελικά απελευθερώθηκε πριν από τρεις ημέρες χάρη στις διαπραγματεύσεις τις οποίες προέβησαν κατά τόπους ηγέτες εκεί υπήρξε μια απαγωγή αλλά το θετικό ήταν ότι οι τοπικοί ηγέτες εκεί ήταν ε, οι οποίοι προέβησαν στη διαπραγμάτευση για την απελευθέρωση αυτού του ατόμου. Άρα λοιπόν σημαντική δουλειά που κάνουμε στην Νότια Λιβύη και θα πρέπει να συνεχιστεί. Τελευταίο τώρα στοιχείο είναι τα δίκτυα διακίνηση ε, Τι αφορά αυτές τις ε, δραστηριότητες ε, ε διακίνηση λαθρομεταναστών στη Λιβύη, παντού βέβαια στη Λιβύη, όχι μόνο στα κέντρα κράτησης. Ε, και διαβάσαμε και όλοι μας αυτά που αναφέρονται ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις εξοδικασίες. Κάνουμε κάτι σε μια χώρα όπου πραγματικά ο σεβασμός ε, των βασικών δικαιωμάτων δεν είναι εγγυημένος. Πρόκειται πάντως για ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να μας απασχολεί. Εδώ χρειαζόμαστε και διεθνή συνεργασία σε αστυνομικό επίπεδο, σε δικαστικό επίπεδο, σε ερευνητικό επίπεδο και αυτό γιατί και έχουν το δίκτυο των επιχειρήσεων τους εντός εισαγωγικών ε, σε διάφορα σημεία και στην Ευρώπη έχουν διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς, άρα ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε αυτή τη λαθρομετανάστευση, αυτά τα δίκτυα στη συγκεκριμένη χώρα, χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία. Αυτό είναι αποτέλεσμα συλλήψει ε, εκείνων ε, οι οποίοι επιβιβάζουν του ανθρώπου στι ελέμβου δεν θα είναι κάτι το αποτελεσματικό. Εκείνο που θα είναι αποτελεσματικό είναι οι δίκτυε που δεν βρίσκονται στη Λιβύη ή στην Τρίπολη Αυτά από την πλευρά μου και είμαι στη διάθεσή σα σε ερωτήσεις. ευχαριστώ πολύ κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Μας ενημερώσατε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Η κυρία Βεριζιά έχει στήσει το λόγο του μεταξύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Ήμουν και εγώ μεταξύ των βουλευτών που στο πλαίσιο τη Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών επεσγέθησαν την τι ε, τα όσα είπατε τα επιβεβαιώνουν και οι δικές μας εμπειρίες. Και εδώ, αλλά και σε άλλους χώρους συζητήσεως Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στη Λιβύη είναι και εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει παράδοση στην ε, μετανάστευση στη Λιβύη και δεν αρχίσουν διάλογο με την κυβέρνηση, λες και υπάρχει με τις αρχές βαρών της Λιβύης, σαν να υπάρχει μια μόνιμη και σταθερή, μια σταθερή κυβέρνηση στη Λιβύη που να Δυσκολεύομαι λοιπόν ε, να αντιληφθώ πώς μπορούμε να συνομιλούμε και να θεωρούμε ότι θα αντιμετωπιστεί με αυτούς τους όρους η κατάσταση ε, των μεταναστών στο μεγαλύτερο βαθμό τους βρίσκονται εκτός του ελέγχου των αποκαλουμένων λιβικών αρχοχρεωμένων να χρησιμοποιούν Λιβίους, οι οποίοι βεβαίως ε, ζουν υπό το δέος των, ε, τον έλεγχό της, αλλά γιατί κάποιες πολιτοφυλακές θα έχουν, πάλι συγχωρήστε μου την έκφραση, ξεπουληθεί στον πλειοδοτούντα, στον πλειοδότη από τα στοιχεία που μας ε, δίνετε να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν να είστε βέβαιοι για τον αριθμό των κρατουμένων σε αυτές τις συνομιλίες. Είναι... Είναι, αντιλαμβάνομαι, σοβαρό στοιχείο Ταυτόχρονα όποιο γνωρίζει την κατάσταση στη Λιβύη αντιλαμβάνεται ότι κανείς δεν ελέγχει πραγματικά την ζώνη αυτή πέραν των τοπικών φυλών και πάλι, συγχωρήστε μου την έκφραση. Και ένα τελευταίο αλλά ερώτημα είναι αυτό της χρηματοδότησης που αφορά και την ε, εμπορία ανθρώπων και ξέρουμε για νομιμοποίηση στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερωτώ λοιπόν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να το αντιμετωπίσει αυτό, γιατί θα πρέπει για να το αντιμετωπίσει να ε, πλήξει τη ρίζα του κακού Ήταν και πολλές ερωτήσεις της κυρίας Βεργιά. Μόνο αν μπορείτε. Αν μου επιτρέπετε πολύ σύντομα δύο διορθώσεις. Πρώτον, από το Δεκέμβριο υπάρχει διεθνές προσωπικό στη Λιβύη και από την Υπατή Αρμοστία και από τα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε ε, την χρήση των ε, συμβαλωμένων ε, υπεργολαβικά όπως θα λέγαμε έναν, ε, χρησιμοποιούμε δηλαδή ένα μηχανισμό που μας επιτρέπει να έχουμε το διεθνές μέρος, ναι, ε, υπάλληλος από το διεθνές προσωπικό ήταν αυτός που απήχθη και για τα κέντρα κράτησης, μια διευκρίνηση, όταν μιλούμε για κέντρα κράτησης, μιλούμε για αυτά που διαχειρίζεται η κυβέρνηση, με ποιον τρόπο συμβαίνει αυτό, ρυθμός ιδιωτικών κέντρων κράτησης, των οποίων ούτε τον αριθμό γνωρίζουμε, ούτε τον αριθμό των κρατουμένων εκεί, ούτε την τοποθεσία. Αλλά ε, δεν περιλαμβάνουμε αυτά τα κέντρα στις συζητήσεις μας, γιατί δεν τις ε, πολιτοφυλακές. Περνούν από το Υπουργείο, σε, ιδιωτικούς, σε ιδιωτικές πολιτικοφυλακές, κάποιοι αξιωματού κέντρα κράτησης. Καθημερινά δουλεύουμε εκεί με το προσωπικό, είναι διεθνές, είναι ε, ντόπιοι και έτσι έχουμε μια καλή εικόνα των ε, κρατουμένων εκεί. Οι επαναπατρισμοί γίνονται από εμά τους ίδιους και η καταγραφή βέβαια ναυλωμένα αεροπλάνα για να τους στείλουμε στα σπίτια τους. Όλα τα άλλα που είπατε, γι' αυτό γνωρίζουμε καλά την κατάσταση, όλα τα άλλα που είπατε βέβαια τα επικυρώνω κι εγώ, είναι σωστά. Από πλευρά Ηνωμένων Εθνών στην Λιβύη παρόντες κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τα δυνά των Λιβύων αλλά και των μεταναστών. Προφανώς και δεν υπάρχει αρχή η οποία να έχει ξεκάθαρα τον έλεγχο ώστε να εξασφαλίσει. Όχι ότι θα αυτή μια συμφωνία, γιατί η συμφωνία έχει τον έλεγχο ενό συγκεκριμένου κομματιού τη επικράτεια, δεν πρόκειται για κεντροκράτη είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι λοιπόν σοβαρό πρόβλημα αυτό. Και ο μόνος τρόπος που μπορέσαμε να βρούμε για να το αντιμετωπίσουμε είναι διαρκώς να διαπραγματευόμαστε με όλους τους παράγοντες εκεί για να υλοποιήσουμε την ανθρωπιστική μας εντολή και αποστολή. Σε ένα βαθμό ε, εγκαθιδρύσει μια επιτροπή διαχείρισης επιτροπών με διάφορους ε, εκπροσώπους, είτε ερετούς είτε προεστούς ε, των τοπικών κοινωνιών και στόχο έχει αυτή η Επιτροπή να λαμβάνει αποκριτηθεί η κοινότητα, είτε πρόκειται για τη διάνοιξη ενός πηγαδιού, ενός δρόμου, ίδρευση, άρδευση, σχολεία κτλ. Κάνουμε μικρό παρεμβάσεις που είναι χρήσιμες για την κοινότητα και τις οποίες έχει επιλέξει η ίδια η κοινότητα, η είναι τοπικό, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να μάθουν να δουλεύουν περισσότερο μαζί. Δηλαδή προσπαθούμε να βελτιώσουμε και την κοινωνική συνοχή της κοινότητας. Αυτή. Ορισμένο ελέγχο που έχει η κυβέρνηση στην επικράτεια της Λιβύης. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν. Είναι πολύ απλό. Την κυβέρνηση Εθνικής Συνένεσης που είναι η μόνη διεθνώ αναγνωρισμένη κυβέρνηση, και προσπαθούμε να του βοηθήσουμε να φέρουν τα αποτελέσματα που μπορούν. Βοηθούμε επίση και στην ε, εκπαίδευση των λιβικών αρχών ε, όσον αφορά ε, στη διαχείριση του ζητήματος της έντυπης μετανάστευσης συμπεριλαμβανομένων των πτυχών των ανθρωπινών δικαιωμάτων που αποτελεί σημαντικό κομμάτι συστατικό στοιχείο όλων όσων κάνουμε σε θέματα έντευσης συμπεριλαμβανομένων των πτυχών των ανθρωπινών δικαιωμάτων που αποτελεί σημαντικό κομμάτι συστατικό στοιχείο όλων όσων κάνουμε σε θέματα οικοδόμησης δυνατοτήτων και κατάρτιση. Αυτό επηρεάζει φυσικά και τα όσα μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η τα στα κέντρα κρατουμένων. Μερικά, όπως είπαμε, είναι εκτός ελέγχου της κυβέρνησης. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, υποχρεούμεθα να τηρούμε και του ε, κανόνε τη ε, κυριαρχία, ε, τη Εθνική Κυριαρχία. Η δουλειά μα το γνωρίζουμε, φέρει μερικά αποτελέσματα. Αυτά μπορούμε να κάνουμε μόνο και ο μόνο τρόπο να επιληθούν όλα αυτά τα ζητήματα είναι η πολιτική σταθεροποίηση τη χωρα Μια ειρηνευτική συμφωνία η οποία θα εγκαθιδρύσει μια αναγνωρισμένη, νομιμοποιημένη κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να διοικήσει αποτελεσματικά τη Λιβική επικράτεια στο σύνολό της με την υποστήριξη ενός ε, ενωμένου στρατού. Αυτό είναι εύκολο να το λέει κανείς εδώ ή οπουδήποτε αλλού και στη Λιβύη ενός ε, ενωμένου στρατού. Αυτό είναι εύκολο να το λέει κανείς εδώ ή οπουδήποτε αλλού ε, και στη Λιβύη τα πολέμησης του ξεπλήματος μαύρου χρήματος Πρώτα απ' όλα με τη διατήρηση μιας ε, ε, λίστας παρακολούθησης των χωρών υψηλών κινδύνου για το ξέπνιμα μαύρου χρήματος και στην επιβολή κυρώσεων σε αυτούς. Αυτή η συζήτηση γίνεται στη Νέα Υόρκη, αλλά πέραν το συζητήσουμε στη δυτική και νότια πλευρά της Λιβύης. Και το τελευταίο θέμα, διεθνές προσωπικό. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα είδατε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται, ταξιδεύει στην Τρίπολη, μία ή δύο φορές τη βδομάδα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, ε, κύριε Πικέ, κύριε Αμπρόσε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Ήταν πολύ λεπτομερής η παρουσιάση και η ενημέρωση. Να ζητώ, προσπαθήστε να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι Ε, ε, από τις παρεμβάσεις και τις απαντήσεις ε, βλέπουμε λίγο μεγαλύτερη ισοδοξία. Βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιος διάλογος και κάποια ελπίδα για το μέλλον. Αλλά όλα αυτά φυσικά υπό όρους. Ε, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα σχέδιο δράσης και όπως φαίνεται θα μπορούσε κανείς να πει ότι διακρίνει ένα φως στο άκρη του τούνελ με τις εκλογές εφόσον υπάρξει η απαραίτητη νομική βάση φυσικά, αλλά στα όσα ακούσαμε από τον κύριο Αμπρόζη, ότι καταφέραμε να ανακόψουμε κάποιες καταστάσεις ε, από τις πιο τραγικές ε, και τη σιγά σιγά καταφέρνουμε να επαναφέρουμε κάποιους εκτοπισμένους στα σπίτια να δημιουργήσουμε ένα, αυτό τον ε, διακοινωτικό διάλογο που είναι απολύτως απαραίτητος για να εγγυηθούμε τη σταθερότητα και μετά και το πρόγραμμα εθελούσες επιστροφής. Ε, ε, όλα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Το μόνο που μένει είναι το ζήτημα, το σημαντικό ζήτημα κατά την άποψή μου του νομοποίησης εσόδων παράνομες δραστηριότητες. Το ξέπλυμα χρήματος για μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αρκεί να βάζουμε χώρε και να τι βγάζουμε από μια λίστα. Στο παρελθόν είχαμε συνεργαστεί με την Ελβετία για να ανοίξουμε, να ταυτοποιήσουμε του λογαριασμού, να βρούμε πού βρίσκονται αυτοί οι πόροι που έχουν μετακινηθεί από το δικτάτορα. Θα έπρεπε κανείς να μπορεί, όταν έχει τη διαδικασία τέτοιου δυνατότητες και πληροφορίε. Δυνατότητε χρήση υπολογιστών θα έπρεπε να μπορούμε να δούμε ποιοι είναι οι, κύριοι πέτοι αυτής της ανθρωπιστικής τραγωδία. Στις διακηρύξει μας λοιπόν, πώς να το πω, θα έπρεπε να κάνουμε μια προσπάθεια στο βαθμό του δυνατού να εμπλέξουμε όλους τους ενδιαφερομένους και όχι να αποφασίζουμε ευθύς εξ αρχής ποιος είναι καλό και ποιος είναι κακός είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε μια προσέγγιση ευρωπαϊκή με όσο το δυνατόν λιγότερους αποκλεισμούς ώστε να μην επαναλαμβάνονται αυτές οι καταστάσεις και να μην προστίθενται ε, πολιτικές αντιπαρθέσεις. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφοι για τις παρουσιάσεις σας. Ισχύει σε ό,τι αφορά τα εν λόγω δεδομένα και τη δραστηριότητα της εν λόγω εταιρείας και ο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπει ότι ένα δικαστήριο τρίτης χώρας ή η αρχή μιας τρίτης χώρας έχει το δικαίωμα να, ε, άμεσης πρόσβασης στη βάση δεδομένων. Όπως ε, προβλέπει και ο κανονισμός, ο γενικός κανονισμός ε, για την προστασία των δεδομένων, πάντοτε χρειάζεται συγκεκριμένη νομικός, ε, νόμιμος τρόπος για πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα είναι μέσω των διεθνών συμφωνιών που ισχύουν μεταξύ ε, Ηνωμένων Πολιτείων αλλά και των κρατών μελών με τις ΗΠΑ. Ζητώ συγγνώμη. Δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε εδώ στην ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ναι, μας αναγκάζει να τα κάνουμε έτσι. Δηλαδή ήρθα τόσο καθυστερημένο γιατί ήμουνα στην ε, διακοινοβουλευτική συνεδρίαση με τις χώρες και μόλις τώρα. Αλλά εν η περιπτώσει ε, είχαμε τη δυνατότητα πριν από μερικές μέρες να ανταλλάξουμε απόξεις με ε, νομικούς οι οποίοι εξειδικεύονται στα ζητήματα ιδιωτικότητας και την ε, μη αμοιβαία αναγνώριση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης από ε, σημαντικούς άλλους εταίρους ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικότερα δε τις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν εδώ έχει προκύψει ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα, δηλαδή μια υπόθεση όπου το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών εξαναγκάζει την Microsoft να διαθέσει δεδομένα τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα εκτός ε, ΗΠΑ και μάλιστα σε μία ευρωπαϊκή χώρα, της Ένωσης δηλαδή, και δεδομένα τα οποία αφορούν ακριβώς την ιδιωτικότητα ε, των πολιτών της ε, Ένωσης. Άρα εδώ λοιπόν θίγονται μια σειρά αποζητήματα για μας ως πολίτες της Ένωσης. Καταρχήν θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία εμείς τα εκπονήσαμε και τα οποία εμεί σεβόμαστε ακριβώ και με την υιοθέτηση του πακέτου, του νομοθετικού πακέτου για την προστασία των δεδομένων. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το ότι έχουμε να κάνουμε εδώ και με ένα ζήτημα διεθνού δικαίου. Δηλαδή εθνικού διεθνού δικαίου, με βάση το οποίο ε, οφείλει κανείς να συμμορφώνεται με την ομοθεσία του κράτους εκείνου όπου ισχύει σε επίπεδο δηλαδή εδαφικής επικράτειας μια συγκεκριμένη νομοθεσία. Η εν λόγω δηλαδή ε, νομοθεσία είναι εκείνη που ισχύει και όχι η νομοθεσία ε, της χώρας εκείνης στην οποία εκδόθηκε για παράδειγμα η άδεια λειτουργίας ή λειτουργία η έδρα της εν λόγω επιχείρησης. Άρα αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι η εν λόγω υπόθεση ε, της Microsoft ενώπιον του Ενωτάτου Δικαστηρίου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ένωση γενικότερα και γι' αυτό θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε προσεκτικά και να αντλήσουμε ε, τα διδάγματα από την απόφαση που θα προκύψει, γιατί ήδη έχουμε αντλήσει κάποια διδάγματα σε ό,τι αφορά τη μη αμοιβαιότητα με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση δεδομένων. Εάν ένας Ευρωπαίος δικαστής δηλαδή προσπαθήσει να αξιώσει τέτοιου είδου δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην επικράτεια των ΗΠΑ, ε, νομίζετε ότι δεν θα πει τίποτα η Αμερικανική πλευρά, θα το επιτρέψει. Δεν νομίζω. Και πάλι δηλαδή, ουσιαστικά το γενικότερο πλαίσιο ε, είναι αυτό των, της αβεβαιότητας ε, που προέκυψε και από τις αποφάσεις του δικαστηρίου σε σχέση με την Διατατική Συμφωνία, με την Συμφωνία και την προστασία των δεδομένων. Ουσιαστικά δηλαδή αναφέρουμε εδώ στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης σε ό,τι αφορά τα ε, ψηφιακά δεδομένα εκεί στην Ελλανδία, που ουσιαστικά απαγόρευσε το ε, γνωστό σε privacy shield. Και μετά τη σχετική απόφαση που συνέχεια κύρωσε και το Safe Harbor, έχει προκύψει πραγματικά μια γενικότερη αβεβαιότητα γιατί ε, αυτά τα νομικά πλαίσια ήταν αποτελεσματικά και είχαν αντίκτυπο στην νομοθεσία ορισμένων κρατομελών. Άρα λοιπόν αυτές οι αβεβαιότητες θα αρχίσουν τώρα να ανακύπτουν, οι επιπτώσεις δηλαδή αυτές οι γενικότερες αβεβαιότητες, οπότε πρέπει και εμείς να προετοιμαστούμε συζητώντας αυτά τα ζητήματα. Ε, Ευχαριστώ. Και το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι πάλι δικό σας κύριε Άλμπρεχτ. Ενίσα.